μας για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ενίσχυση του ρόλου μας στην περιοχή αλλά και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία εν ώψη της μελλοντικής της ένταξης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια φυσική συνέχεια με το Μηχανισμό Πρωταξιακής Βοήθειας 2, τον οποίο πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα υποψήφια κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κιουτσούκ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Σόλτες για τους ε, πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό που παρέχει πρενταξιακή βοήθεια, πολύ αποτελεσματικό και στο μέλλον και απολύτως απαραίτητο. Η τρίτη γενιά του μηχανισμού πρωταξιακής βοήθειας δράζεται σε νέε αρχές ε, με τις οποίες συμφωνούμε. Αυτή η νέα προσέγγιση ε, βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων στη χρήση των κονδυλίων ε, είναι θετική και θα ε, επιτρέψει μια πιο χρηστή διαχείριση των κονδυλίων και θα αυξήσει και την αποτελεσματικότητα. Έχω κάποια σχόλια πάντως. Μέχρι στιγμή, οι υποψήφιε για ένταξη χώρε είχαν προγράμματα με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους από τα δύο πρώτα προγράμματα πρωταξιακή βοήθειας. Θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέε αρχέ του τρίτου μηχανισμού πρωταξιακή βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσγειωμένοι ρεαλιστές και να αφιερώσουμε κονδύλια στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην ευαισθητοποίηση των υποψηφίων χωρών για τις νέες αρχές προκειμένου και ο τρίτος μηχανισμός προταξιακής βοήθειας να υλοποιήσει του στόχου του. Το ενδιαφέρον ε, με τη νέα προσέγγιση είναι ότι περιλαμβάνουμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν πολλά να προσφέρουν, έχουν πλούσια πείρα και μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση των νέων κονδυλίων. Επίσης, με τη νέα προσέγγιση θα έχουμε διευκόλυνση της περιφερειακής συνεργασίας, που είναι εξαιρετική ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, το λόγο ο κύριος Γιάρομιρ Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το 2015 είχαμε την ενδιάμεση στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διεύρυνση που περιλαμβάνει όλες τι χώρε των Δυτικών ε, Βαλκανίων που πήραν το καθεστώ υποψήφια χώρας και συνεχίζει το διάλογο με τις ε, ε, χώρε αυτές. Η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί και στα πλαίσια του νέου μηχανισμού προταξιακή βοήθεια, του τρίτου μηχανισμού Προταξιακή βοήθεια, που στόχο έχει να βελτιστοποιήσει το θετικό αντίκτυπο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δίνεται έμφαση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ε, σταθερά, θεσμι... σταθερά θεσμικά όργανα, κράτος δικαίου, προστασία μειονοτήτων και στην ικανότητα να αναπτύξουν οι ψήφιες χώρες ανθεκτικότητα στον ανταγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 14,5 δισεκατομμύρια ε, είναι ο προϋπολογισμός για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού ε, κάτι που είναι αντίστοιχο με την ετήσια συνεισφορά της Τσεχίας στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Επίσης, ε, έχουμε στόχους όπως η μετανάστευση, καινοτομία, προστασία του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών, προγράμματος έρασμος ΣΥΝ λοιπά. Επίσης θα πρέπει να ελεγχθούν εξουσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση αξι... αντικειμενικά κριτήρια. Πάντως το... η ομάδα μου δεν μπορεί να δεχθεί την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Τώρα για το EFDD ο κύριος Κάρβερ. Ε, πρόκειται μάλλον για την τελευταία μου ομιλία εδώ μέσα και πραγματικά παρακολουθώ την τεράστια απογοήτευση που επικρατεί τα τελευταία πέντε χρόνια παρά τις ε, διαφωνίες σας συνεχίζετε στην ίδια κατεύθυνση προς όλο ένα και στενότερη ένωση χωρίς να παρατηρείτε την πραγματικότητα γύρω σας. Δείτε την Τουρκία παραδείγματο ε, χάρη. Ε, είχαμε μια έκθεση αυτόν τον μήνα που μας λέει ότι υπάρχει υπαναχώρηση στα θεμελιώδη δικαιώματα και όμως επιμένετε να δώσετε λεφτά στον κύριο Ερντογάν την ίδια στιγμή που δεν αναγνωρίζετε την ασυμβατότητα, ούτε τη λέξη δεν μπορώ να πω, με τις θεμελιώδε σα αξίες. Ε, και ασκείτε όμως κριτική στη Ουγγαρία και Πολωνία. Μα δεν βλέπετε την υποκρισία σας. Πόση ζημιά πρέπει να κάνετε πριν αντιληφθείτε το ότι δεν εκπροσωπείτε τι ανησυχίες των πολιτών σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω τώρα έχει ο κύριος Μποργέτσι από το Κυρία Πρόεδρε, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και αναφερθήκαμε και στο ζήτημα της Τουρκίας. Εγώ θα ήθελα να αφαιρθώ όμως σε μια άλλη περίπτωση που πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε τελικά και αν θα πρέπει τελικά να παρέχουμε προταξιακή βοήθεια. Πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρούμε ότι έχουμε διακριτική μεταχείριση της σερβικής μειονότητας ε, από, την, από το 2000 το 2004 στο Κωσυφοπαίδιο. Νομίζω ότι πέρα από την αστολή της προταξιακής βοήθειας που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο πιο επισταμένα με την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να προωθούμε εμεί κάποιε αξίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη να υπάρχει μια σαφή διακριτική μεταχείριση. Και α μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών που επιβεβαιώνουν μια τέτοια πολιτική διακριτική μεταχείρισης που στρέφεται κατά των ίδιων των Σέρβων τη σερβική μειονότητα στο Κωσφοπέδιο, άνθρωποι οι οποίοι ζουν εντελώς παραγωνισμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα βασικά του δικαιώματα και ούτε καν το θρησκευμά του, το ορθόδοξο θρησκευμά του. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπορκέζιο. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ντέβιτ Μακάλιστερ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη ακούσαμε, το μέσο αυτό παραμένει το κυριότερο μέσο για να βοηθήσουμε τον μετασχηματισμό των χωρών αυτών που στόχο έχουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως η τρίτη γενιά αυτού του μέσου από το 2021 μέχρι το 2027 θα εξυγχρονιστεί για να αντικατοπτρίζει τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται εξτάμενα προγράμματα. Είναι καλοδεχούμενο αυτό. Το ότι δηλαδή στην έκθεση αυτή ζητάμε μια αποτελεσματική αρχή για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ζητάμε μια αυξημένη αίρεσιμότητα και τη δυνατότητα αναστολής της κοινωτικής χρηματοδότησης ε, στην περίπτωση αδυναμίας σεβασμού των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους εισηγητές. Είναι πράγματι κάτι το σωστό. Σας ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ. Ο κυρία Τζούλι μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας. Παίζει πράγματι έναν σημαντικό ρόλο στην εξωτερική μας ε, πολιτική με τις χώρες της διεύρυνσης και θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προωθήσουμε τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στις ε, χώρες αυτές, ανθρώπινα δικαιώματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρέπει να είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Και έχουμε εδώ πέρα μια ευελιξία που θα αποδειχθεί πολύ σημαντική στη σχέση μας με την Τουρκία. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να προσαρμόσουμε την πολιτική μας αυτή και να εστιάσουμε στην κοινωνία των πολιτών αντί για τις κρατικές υπηρεσίες. Και βεβαίως είμαι πεπισμένος εγώ παρά τα όσα κάνει ο κ. Ερντογάν πως χώρα αυτή ανήκει στην Ευρώπη. Οι επαφές μου με την τουρκική κοινωνία των πολιτών με έχουν πείσει πως οι Τούρκοι πολίτες θέλουν ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία και να είναι μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και όσον αφορά τα Βαλκάνια, πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ε, την οικοδόμηση θεσμών και την κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γουόρντ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Καστάλντο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω εδώ πέρα πραγματικά ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερο και επιβεβαιώνεται και στη σημερινή συζήτηση. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορώ να μιλήσω με απόσταση, αν θέλετε, με ψυχρότητα, όσον αφορά τις τεχνικές πλευρές ε, του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας, νομίζω θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τους στόχους του μηχανισμού αυτού. Στα πλαίσια του υπα 3 θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη προσαρμογή στην πολιτική κατάσταση των εταίρων μας. Χάρη στην εξαιρετική εργασία που έχουν κάνει οι συνάδελφοι Σαλαφράκα και Φλέκενστάιν, αυτό όντως θα πρέπει να συμβεί μέσω από την πρόταση αυτή. Νομίζω πραγματικά ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για τον προγραμματισμό, την κατάρτιση του μηχανισμού αυτού και την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού. Και μπορεί το Κοινοβούλιο επίση να έχει και το δημοκρατικό έλεγχο για αυτό το μηχανισμό. Επίση, είναι πολύ θετικό και αναγκαίο παράλληλα, θα έλεγα, το να ενισχυθεί η προτινόμενη αιρεσιμότητα και να έχουμε εκταμείευση των κονδυλίων βάσει των επιδόσεων και συγκεκριμένων σημείων συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά τι επιδόσει των, κρατών, των εταίρων κρατών και θα πρέπει μάλιστα να προβλέπεται και αναστολή των, της χρηματοδότης κάθε φορά που έχουμε οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπεχάγης και ιδίω όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως αυτά τα σημεία αναφοράς και θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε και στην Τουρκία η οποία χάνει όλο και περισσότερο την αξιοπιστία της. Κυρίε και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθούμε τι βασικέ αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη πολιτική διεύρυνση. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε να έχουμε τον ξεχωριστό αυτομηχανισμό ακόμα και την περίοδο αυτή που προσπαθούμε να θεσπίσουμε και έναν ενιαίο μηχανισμό γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε το μηχανισμό αυτό αύριο, να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά των προηγούμενων ετών. Χάρη στο νέο αυτό μηχανισμό προταξιακή βοήθεια, θα έχουμε ένα πολύ θετικό εργαλείο στα χέρια μα που θα δεσμεύσει όχι μόνο τι χώρε εταίρου, αλλά και εμά του ίδιου για να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό αυτό πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Άνεμαντς από το ΙΕΝΕΦ. Συναδελφοί, το κοινοβούλιο αυτό ε, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει το όνειρο κάποιον ότι θα γίνει κάποτε κράτος μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να σταματήσει και την ροή δισεκατομμυρίων. Έχουμε 140.000 άτομα στην ε, φυλακή, μεταξύ των οποίων χιλιάδες ε, ε, δίκαστες ε, οι οποίοι απολύθηκαν 150 ε, μήμοι έχουν κλείσει εκατοντάδες δημοσιογράφοι έχουν απολυθεί και συλληφθεί. Αν το διαβάσει αυτό κανείς σε συνδυασμό με τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία επενδύει στην υπηρεσία θρησκευτικών υποθέσεων για να χτίζει τζαμιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία Δηλαδή χρηματοδοτούμε την Τουρκία για να χτίζει εδώ πέρα τζαμιά. Ε, σας παρακαλώ να σταματήσετε αμέσως αυτήν την χρηματοδότηση. Δεν έχει κανένα νόημα και δεν θα ενταχθεί ποτέ αυτή η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Άνεμαν. Ο Έντουαρτ Κούκαν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ του δύο συνεισηγητέ. Ε, συγχαρητήρια για το εξαιρετικό του έργο. Συγγνώμη κύριε Κούκαν Μία μπλε κάρτα έχει σηκωθεί για τον κύριο Άνεμανς. Δέχεται την ερώτηση με την μπλε κάρτα, κύριε Άνεμανς. Ναι, ο κύριος Φλέκερσταϊν μισό λεπτό παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Φλέκενστάιν. Κύριε Άνεμανς, δεν ακούτε τι λέμε πριν από λίγες εβδομάδες αποφασίσαμε αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είπαμε ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση στην κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία. Με το μηχανισμό Πενταξιακής βοήθειας 3 έχουμε ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να πούμε αν δεν λειτουργεί ε, έχουμε και λιγότερα λεφτά. Πηγαίνουμε λοιπόν προς σωστή κατεύθυνση. Ε, τι μας λέτε τα ίδια και τα ίδια. Ε, νομίζω ότι πλέον δεν έχουν νόημα. Έχω άδικο. Ε, έχετε τον λόγο κύριε Άνεμανς για να απαντήσετε. Κύριε Φλέκενσταν, με κάθε σεβασμό η συζήτηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ενός μηχανισμού ο οποίο δεν έχει νόημα. Η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και δεν θα γίνει. Μα δεν ζητάω πόλεμο με την Τουρκία. Θέλω καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτό το όνειρο περί ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, έτσι. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κούκαν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εκτιμώ ιδιαίτερο στο άρτιο πόνημα των δύο συνεισηγητών. Συγχαρητήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε επενδύσει σχεδίων και προγραμμάτων που στόχο έχουν την προώθηση του κράτους δικαίου, τη λειτουργία των, των δημοκρατικών θεσμών και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, Συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθεροτυπία ή τη ελευθερία των ΜΜΕ. Για να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι είναι απαραίτητη συνεργασία και με τις κυβερνήσεις αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, την οποία θα, την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε ενεργά. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα κονδύλια μας και τη χρηματοδότηση προς την περιοχή με, σοφ... συνετό τρόπο, γιατί είμαστε μεγαλύτερος δωρητής και μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος όλων των χωρών της περιοχής. Επενδύουμε σε υποδομές, σε ενεργειακά δίκτυα, στο περιβάλλον, στη γεωργία, στα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε αναμένουμε από τις χώρες αυτές να λάβουν ε, σοβαρές δεσμεύσεις για ε, μεταρρυθμίσεις ε, και για σεβασμό των θεμελιωδών αξιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κούκαν. Το λόγο κυρία Νίνα Γκίλ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια και στους δύο εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν ενώ καλωσορίζω τα γενικά σχέδια της Κομισιόν για περισσότερες επενδύσεις στην εξωτερική δράση στο νέο πι δελταπί με κάπως επιφυλακτική για την αύξηση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας. Εγώ είχα πάει με την Επιτροπή Εξωτερικών στις χώρες αυτές. Αυτό το οποίο μου προξενεί έκπληξη πάντα είναι ή μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης της χρηματοδότησης σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Οπότε οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Πρώτον, κύριε Χάν, με ακούτε. Ε, η DG NIR, η Γενική Διεύθυνση Γειτονίας, πώς εκτιμά την ικανότητα απορρόφησης των χωρών αυτών, το λαμβάνει υπόψη. Δεύτερον, μόλις ακούσαμε πώς το Κοινοβούλιο ψήφισε να ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, δεδομένου του ότι είναι μακράν ο ε, μεγαλύτερος δικαιούχος κονδυλίων, πώς θα επηρεαστεί η εκταμίευση και τρίτον, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, η αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία δεν είναι και η καλύτερη. Ανταυτού ε, χαίρονται και υπερτιμούν ιδιαίτερως τις επενδύσεις της Ρωσίας και της Κίνας. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκίλ, τον λόγο έχει ο κ. Τσόκα. Απευθύνομαι στις αλβανικές αρχές. Σε αυτές θα ήθελα να αφαιρθώ και σαφώς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη χώρα αυτή στα πλαίσια του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας, ενώ έχουμε οι οικογένειες αλβανικές οι οποίες απειλούν τους συμπολίτε μας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν απειλέ, συγκεκριμένε απειλέ, απειλές οι οποίες γίνανε από μια αλβανική οικογένεια προς τον Φραντσέσκο Τσιτσινιάνο, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν από μερικές ε, μέρες. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η οικογένεια αυτή πιστεύει ότι μπορεί εκβιάζοντας την οικογένεια του ταλού αυτού πολίτη να καταφέρει να πάρει λίτρα, ουσιαστικά να καταφέρει να εκφοβήσει την οικογένεια κατά αυτόν τον τρόπο. Τέτοια φαινόμενα όμως έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή δημιουργούνται εγκληματικές ομάδες πραγματικές οι οποίες στρέφονται κατά τον ίδιο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το πρόβλημα το βασικό που έχουμε είναι ότι χρηματοδοτούμε τελικά τους υπεύθυνους για τις πράξεις αυτές αντί να πρημοδοτούμε τους έντιμους πολίτες. Ο κύριος Πέτερλ έχει το λόγο. Ε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο μηχανισμό προταξιακή βοήθεια είναι ένα τρόπο να βοηθήσουμε τι υποψήφιε για ένταξη χώρε στην ενταξιακή του πορεία. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βελτιώσει το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Θεωρώ ότι η υποψηφιότητα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα είναι βασικό βήμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το σχέδιο ειρήνης μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί όσο το ε, μένουν τα Δυτικά Βαλκάνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτές τις χώρες για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις ευρωπαϊκές πολιτικές και μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από του βασικού τομεί στου οποίου θα πρέπει να επικεντρώνεται ο μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια είναι η δημιουργία θεσμικών οργάνων, η πάταξη τη διαφθορά και η η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών φορέων, βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ε, θεσμούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρικιέν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την αρτιότατη εκθεσή τους. Ο μηχανισμός πρωταξιακής βοήθειας είναι δισεκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα μία επένδυση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταστήσουμε έτσι πιο ευημερή και πιο ασφαλή την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζοντα τη σταθερότητα και την ευημερία των γειτονικών μα χωρών, των στενότερων γειτόνων μα, στηρίζοντά του στην πρωταξιακή του πορεία. Η διαδικασία διεύρυνση δίνει μια όθηση στην οικονομική ολοκλήρωση των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι συμφωνίε με τι χώρε τη διεύρυνση, η απελευθέρωση του ε, εμπορίου είναι πολύ σημαντική. Και ο μηχανισμό προταξιακή βοήθεια τρίτη γενιά στηρίζει τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και τη Τουρκία κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την πάταξη τη διαφθορά, για την προώθηση τη οικονομική ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία τη οικονομία αγορά, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα. Στηρίζοντας λοιπόν τους γειτονές μας στην πρωταξιακή τους πορεία, η αιρεσιμότητα του μηχανισμού πρωταξιακής βοήθειας επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα αναστολή σε περίπτωση παραβίασης των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι σαφής και αυτή η δυνατότητα αναστολής να στέλνει ένα χειρό μήνυμα προς τις υποψήφιες χώρες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η επόμενη ομιλήτρια, που είναι η τελευταία ομιλήτρια στη συζήτηση αυτή, η κυρία Ζέλιανα Ζόφκο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, δύσκολη καιρή και για τις ε, υποψήφιες για ένταξη χώρες και δεδομένου αυτής της αντικσότητας θα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη τη στήριξη των χωρών αυτών και στον τρίτο μηχανισμό προταξιακή βοήθεια και να επικεντρωθούμε σε μέτρα που δημιουργούν ε, ενίσχυση των εκατομμύτων ασφάλεια ε, και τη αθεκτικότητα των θεσμών. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία για το μηχανισμό προταξιακή βοήθεια είναι ένα στρατηγικό σχέδιο πρόθεση και επικοινωνία. Με τι τροπολογίε μου επισημαίνω ότι μόνο με την καλύτερη προβολή αυτού του μηχανισμού και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες θα, βελτιω... θα βελτιστοποιήσουμε το βασικό μας μηχανισμό για τη σταθερότητα και η ειρήνη στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζόφκο. Περνάμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Έναν ομιλητή έχω μόνο σε αυτή τη διαδικασία που είναι ο κύριος Στάνισλαφ Πόλτσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πιστεύω ότι ε, οι χώρες αυτές, οι οποίες θα ήθελαν κάποια στιγμή να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συνειδητοποιούν ότι τις υποστηρίζουμε. Θα πρέπει να το βλέπουν αυτό ξεκάθαρα. Και τα όσα λέω σχετίζονται και με την όλη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο για την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στι χώρε αυτέ στα πλαίσια του μηχανισμού προταξιακή βοήθεια, να κινητοποιήσουμε συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει στι χώρε αυτέ. Παράλληλα, χαιρετίζω την πρόταση που γίνεται στην έκθεση αυτή να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των κατεξοδότηση πράξεων. Όσον αφορά τώρα την Τουρκία και την προταξιακή βοήθεια προς τη χώρα αυτή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι Τούρκοι πολίτες να αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποστηρίζει. Κατά την άποψή μου όμως η Τουρκία, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν είναι καθόλου έτοιμη να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι Επισμένει ότι αυτό άλλωστε πιστεύει και η τουρκική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα διάλογο πάντως με τη χώρα αυτή. Υπάρχει σημαντική παραβίαση βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα με τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Ελπίζω να προσέξατε ότι η κυρία Γκέλη έκανε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο κυρία και άλλοι συναδελφοί σας. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή. Το συμπέρασμά μου είναι ότι έχουμε πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε και αναμένουμε την επικοδομητική συνεργασία μας και υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία στο ότι θα πρέπει να διατηρηθούν κάποιες παραμετρικλίδια. κλειδιά. Έχουμε λοιπόν μια σύνδεση θεμελιωδών δικαιωμάτων και κρατσοκαίου με τους άλλου τομεί της ένταξης, δηλαδή οικονομική διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσει. η ενίσχυση της δημόσιας διοίκηση και των δημοκρατικών θεσμών βεβαίως θα συνεχίσουν να αποτελούν το κύριο θέμα της συνεργασία μας. Επίσης βεβαίως και ο συντονισμό της διασυνοριακή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις ε, χώρες δικαιούχους που είναι πολύ πιο σημαντική στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα δεν αφήνουμε την Τουρκία μόνη τη. Ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε σημαντική στήριξη για να στηρίξουμε, όπως είπε ο κ. Φλέκενστάιν, την δημοκρατική διαδικασία και την κοινωνία των πολιτών. Είναι αυτή η δυναμική, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Τουρκία και να προσαρμοστούμε στην ε, κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται ε, στις ε, σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Και έρχομαι τώρα σε κάποια σχόλια της κυρίας Μάλετιτς αλλά και κάποιες ανησυχίες της κυρίας Γκίλ. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Γι' αυτό θα ήθελα να εστιάσω σε μια καινοτομία, το ότι έχουμε μια πιο στρατηγική εστίαση που μας επιτρέπει να ανταμείψουμε την πρόοδο και να αυξήσουμε και την ευελιξία για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των εταίρων μας. Κάτι το οποίο σημαίνει πράγματι ότι εάν υπάρχουν προβλήματα στην ικανότητα απορρόφησης στο μέλλον μπορούμε και να τα αποφύγουμε με το να εστιάζουμε στις θεματικές προτεραιότητες. Και κάποιος είπε ότι ίσως υπάρχουν προβλήματα στη χύψη χώρα στο να ετοιμάσει όριμα έργα. Η εμπειρία μας, εντάξει, δείχνει ότι πάντα είναι έτοιμες να προετοιμάσουν κάποια έργα, αλλά καμιά φορά στην χή στον χ θεματικό τομέα, άλλες φορές σε άλλους. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για να προετοιμάζουμε έργα με έναν τρόπο που να μπορούμε τελικά να τα στηρίξουμε οικονομικά. Αλλά το σκεπτικό των θεματικών προτεραιοτήτων είναι να υπάρχει, θα έλεγα, κάποιο είδους ανταγωνισμός ε, μεταξύ των χωρών αυτών και να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία. Οπότε αν μια χώρα έχει ρίξει περισσότερο βάρος στο κράτος δικαίου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επενδύσει περισσότερα εκεί. Άλλες μπορεί να έχουν εστιάσει περισσότερο στις μεταφορές. Ε, τελικά όμως θα πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρουν την έγκριση, θα λέγαμε, των κρατών μελών ε, για να γίνουν κράτη-μέλη. Αλλά για να φτάσουμε εκεί νομίζω πως καλό είναι να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Βεβαίως, κυρία Μάλετιτς, θα υπάρξουν οι ενδεικτικοί φάκελοι αναχώρα, αλλά βασιζόμαστε στις θεματικές προτεραιότητες και είμαστε πεπισμένοι, όπως είπαν και οι περισσότεροι συναδελφοί σας, ότι αυτό μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, με περισσότερη ευελιξία και να ε, εξυπηρετούμε τα κοινά μας συμφέροντα για να προετοιμάσουμε τις χώρες αυτές, ε, ελπίζουμε, για μια γρηγορότερη ένταξη από ό,τι ε, φαίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι που μας βοηθήσατε για να ξεκινήσουμε με αυτό το πρόγραμμα 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης. Ε, όπως σας είπα, είτε θα κάνουμε εξαγωγή σταθερότητας, είτε εισαγωγή αστάθειας. Και ε, νομίζω πως αυτά τα οποία έχουμε υποβάλει συνεισφέρουν σε αυτόν τον στόχο και σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και αναμένω τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο συνεισηγητές. Πρώτα στον κύριο Σαλαφράνκα. Όπως είπα και πριν, ε, και το τόνισε και ο κύριος Φλέκης στη δικιά του, είναι σημαντικό οι αρχές που διέπουν τον κανονισμό και είναι η βάση της ε, ευρωπαϊκής δράσης. Είναι η ειρήνη, η επανασυμφιλίωση, η ομόνια. Αυτά θα είναι τα βασικά στοιχεία και των μελλοντικών μας εξωτερικών δράσεων, ώστε τα παιδιά που γεννιόνται σήμερα στα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα, να πρέπει να πάνε στη βιβλιοθήκη, να διαβάσουν ε, βιβλία ιστορίας για να γνωρίσουν την αιματοχημένη ε, πραγματικότητα, την ε, αιμοσταγή ιστορία. Και όπως είπε και ο Φλέκενστάιν, ο κύριος Φλέκενστάιν, συνεισηγητής έκθεσης, η έκθεση πραγματικά σηματοδοτεί πολύ μεγάλη πρόοδο και ελπίζω να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, κύριε Επίτροπε, σημειώσαμε την ανάγκη συνοχής μεταξύ τη εξωτερικής πολιτικής μας και τη πολιτική διεύρυνση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ήθελα να τονίσω ότι είμαστε στη διάθεσή σα για να συνεχίσουμε την πρόοδο μα στα θέματα αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία σύμπτωση και κοινέ απόψει και γι' αυτό μπορούμε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε ένα νέο κανονισμό για να αντιμετωπίσουμε τι νέε προκλήσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο εσωτερικά ε, και το, με τα προβλήματα που έχουμε με τον Brexit, να ασχοληθούμε και με τι γειτονικέ μα χώρε που είναι υποψήφιε για ένταξη χώρε και να εμπεδοθούν αυτέ οι σχέσει, να εδραιωθούν σε ένα χρηματοδοτικό μέσο, στο τρίτο μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια. Έχουμε πολλές άλλωστε κοινέ διατάξεις ε, με το μηχανισμό χρηματοδότησης γειτονία ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας και είμαι βέβαιος κύριε Επίτροπε ότι θα βρούμε τρόπους ώστε πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε οριστικοποίηση του κανονισμού για να αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό και με σεβασμό των ε, αξιών και αρχών που σας ανέφερα τις προκλήσεις που έχουμε στην ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαλαφράγκα και τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο εισηγητή που είναι ο κύριος Φλέκενστάιν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις παρατηρήσεις μόνο στο τέλος. Καταρχήν, κύριε Επίτροπε, ε, δεν θέλουμε να υπάρξει σύγχυση μεταξύ των αρμοδιοτήτων, ούτε θέλουμε καμία αλλαγή αλλά θέλουμε να υπάρξει ε, ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ πολιτικής διεύρυνσης ε, και εξωτερικής ε, πολιτικής. Ε, δεν θέλουμε να αλλάξει κάτι ουσιαστικά και πολιτικής γειτονία. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να είναι απολύτως ικανοποιημένοι μαζί μας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διασπείρουμε τα κονδύλια μας εις πλάτος αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα όπως η κλιματική προστασία ε, τα κοινωνικά ζητήματα, η οικονομία, οι θέσεις ε, απασχόλησης. Το ζητούμενο είναι να προσπαθήσουμε ε, σε εξατομικευμένη βάση να κάνουμε κάποιοι περισσότεροι και κάποιοι λιγότερα όποιος ε, καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια θα πρέπει να λάβει από μας μεγαλύτερη μικρότερη υποστήριξη. Και το τελευταίο σημείο, ε, Πρόκειται εδώ για μια, ένα χειρό μήνυμα προς τους ε, πολίτες των περιοχών αυτών. Ανεξάρτητα από την διαμόρφωση του προπολογισμού, ανεξάρτητα από την διαμόρφωση των πλειοψηφών στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα σταθεί πάντοτε στο πλευρό των φίλων μας στα Δυτικά Βαλκάνια και θα προσπαθήσει με τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ να παράσχει ουσιαστική βοήθεια ούτως ώστε να είναι δυνατόν να υπάρξει μια συγχώνευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί και ελπίζω και ότι οι διάδοχοί μας την επόμενη θητεία θα πράξουν το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την κατάσταση στην Αλγερία. Ε, πρώτος θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος κύριος ε, Χάν. Παρακαλώ κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκινώντας από τις 22 Φεβρουαρίου, βλέπουμε μια νέα δυναμική στην Αλγερία με μαζικές διαδηλώσεις ε, μετά και την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Βουτεφλίκα θα κατέβει για πέμπτη φορά στις εκλογές που αρχικά προβλέπονταν για τις 15 Απριλίου. Έκτοτε, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν ουσιαστικά καθημερινά και έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και ο κόσμος ζητάει την απόσυρση του Πετεφλίκα αλλά και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις και του εκλογικού συστήματος. Είναι ειρηνικέ διαδηλώσει σε μεγάλο βαθμό και αντίστοιχη είναι και η στάση των ε, ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαβούλευση και να ακούσουμε τον ε, κόσμο σε ό,τι αφορά την εισαγωγή νέων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Η Αλγερία είναι βασικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, σημαντικά οικονομικά πολιτικά συμφέροντα και δεσμούς που ενώνουν τους λαούς μας. Δεν θέλουμε να υπάρξει αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Οι διμερείς μας σχέσεις τα τελευταία χρόνια κινούνται θετικά και θέλουμε και περιμένουμε να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση. Στι 7 Μαρτίου μάλιστα συναντηθήκαμε και στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε ε, με τον ε, νέο Πρωθυπουργό. Οι διαδηλώσει μέχρι τώρα λοιπόν ήταν ειρηνικέ και η ανταπόκριση των ε, υπηρεσιών ασφαλείας είναι ιδιαίτερα μετριοπαθή. Αυτό είναι θετικό και θα πρέπει να συνεχιστεί. Όπως ξέρετε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ρευστή αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε το του σύνεγγυς ε, και τις σημερινές εξελίξεις. Πρέπει να υπάρξει θετική ε, αντίδραση στις ε, φιλοδοξίες του λαού. Πια πιο ανοιχτή προσέγγιση με περισσότερες ευκαιρίες και σε οικονομικό επίπεδο, ιδίω για τους νέους. Όλες οι εξελίξεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και να συμπεριλαμβάνεται και ο λαός. Οι ίδιοι Αλγερινοί λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους και πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Από τη δική μας πλευρά εμείς ε, ενθαρρύνουμε ε, ελεύθερες, ε, δίκαιες και χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς εκλογές σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει και είναι διατεθειμένη μάλλον να στηρίξει και με τεχνική τεχνογνωσία την εκλογική διαδικασία και με αποστολή εκλογικών παρατηρητών. Βεβαίω, αν το ζητήσει η Αλγερία και αν ε, ε, πληρούνται όλες οι προποθέσεις μιας τέτοιας διαδικασίας. Στηρίζουμε την έκκληση για μια ευρύτερη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και μετάβασης και έχουμε και το σχετικό βήμα ε, για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, αρκεί να είναι μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί γρήγορα πρόοδος Κατανοούμε ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει βούληση ε, να, βρεθεί, ε, να βρεθούν τα απαραίτητα βήματα για το μέλλον. Όλα αυτά θα πρέπει να αποκρισταλωθούν στην πράξη σε μια ομαλή μετάβαση για να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής ε, αυτής της διαδικασίας. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να ακουστεί η βούληση του αλγερινού λαού. Και όπω είπα προηγουμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεθειμένη να συνδράμει την Αλγερία σε αυτή τη διαδικασία, εάν το ζητήσει η Αλγερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Αλγερία στις κοινωνικοοικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις τη, ε, προκειμένου να ακουστεί η βούληση ε, του λαού της Αλγερίας, ιδίως των νέων. Πάντα βέβαια με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας της Αλγερίας και σε ένα πνεύμα εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται και από την πολιτική γειτονία μας. Τα γεγονότα του τελευταίου μήνα έχουν δοκιμάσει την πολιτική οριμότητα στην Αλγερία και περιμένουμε πραγματικά ε, να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Χάν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Πρέντα από το ΕΛΚ. Χιλιάδες ε, διαδηλωτές ε, βρίσκονται στους δρόμους της Αλγερίας κάθε Παρασκευή και ζητούν πολιτική μετάβαση και την απόσυρση του Πρόεδρου Πουτεκλίκ, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να κυβερνήσει τη χώρα. Εδώ και καιρό, δυστυχώς, οι αρχές δεν φαίνεται να ακούνε το λαό, καθώς δεν ε, προτείνουν λύσεις. Η... Στις 28 Απριλίου έλυγε η θητεία του Πρόεδρου, όμως ε, παρατάθηκε. Ε, η εθνική διάσκεψη προτείνεται από την κυβέρνηση απορρίφθηκε από την αντιπολιτεύση και την κοινωνία των πολιτών και από την εξουσία λιποτακτούν ε, πάρα πολύ και ε, το Γενικό Επιτελείο του Στρατού στέλνει αντιφατικά μηνύματα και το είδαμε και σήμερα το απόγευμα η εθνική στροφή των αρχών της Αλγερίας για να καθησυχάσουν τους εταίρους τας ε, ότι μπορούν να διαχειριστούν την κρίση δείχνει την αποτυχία της μετάβασης προτείνει η οικογένεια Μπουτεφλίκα. Η Αλγερία είναι σε διέξοδο, πρόκειται για έναν ε, μεγάλο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγγυάται την περιφερειακή σταθερότητα, η οποία θα ε, μπορούσε ε, να διατηρηθεί αν υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης διαφανές. Οι Αλγερινοί θα περιμένουν την αλλαγή, όμως θα πρέπει να καταπολεμηθεί ριζικά το σημερινό σύστημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάνη για τα λόγια του. Συμφωνούμε και στις ε, ειρηνικές ε, διαδηλώσεις ε, βλέπουμε ότι είναι γεμάτες περηφάνεια και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα για μια βαθιά αλλαγή που να οδηγήσει σε δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές σε ένα εύλογο διάστημα. Συμφωνούμε απόλυτα στο να υποστηρίξουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο και στο να διατηρήσουμε την απαραίτητη υποστήριξη για μια χώρα όπως η Αλγερία, όπου έχουμε μακρά παράδοση σχέσεων. Και χρειαζόμαστε να την κρατήσουμε κοντά και σε αυτή τη σχέση. Επίσης, ε, σε αυτή τη τελευταία θητεία πετύχαμε κάτι που θέλαμε πολύ καιρό, δηλαδή να υπάρξει μια διμερής αντιπροσωπεία μεταξύ Κοινοβουλίου και Αλγερίας εδώ στο Κοινοβούλιο που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και προσφέρουμε και τη δική μας βοήθεια στην Κομισιόν προκειμένου να ε, μπορέσουμε να προωθήσουμε μια ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία. Ευχαριστώ την κυρία Αγία Σέντερ. Μπέλντερ από το ΕΣΥΑΡ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε αδρές γραμμές, στην Αλγερία βλέπουμε ότι υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη για την εθνική κυριαρχία και αυτό έχει ως ε, ε, προέκταση μια μεγάλη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις ξένες επιρροές ε, στη χώρα. Επομένως, καλό είναι να ακολουθήσετε την προσεκτική προσέγγιση που αναφέρατε κι εσείς, γιατί είναι πολύ σύνθετη η κοινωνική κατάσταση στην Αλγερία καθότι έχουμε εδώ και εβδομάδες σε πολύ μαζικές διαδηλώσεις. Από το παλιό δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι νέο. Παρόλα αυτά, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις εκλογές και κατά πόσο ε, θα πετύχουμε ε, τους στόχους που θέλουμε για να πληρωθούν οι φιλοδοξίες του Αργενού λαού. Η Αραβική Άνοιξη του 2011 μας έδειξε ότι η συνέχιση ε, της ε, της ε, αστάθειας φέρνει στο προσκήνιο διάφορες ομάδες οι οποίες τελικά οδηγούν σε περισσότερη αστάθεια. Είναι κάτι Πολύ σημαντικό λοιπόν από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό είναι να υπάρχει ανεξιθρησκεία για όλου ε, του Αλγερινού και να προσέχουμε του φανταμεταλιστέ από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από την άλλη, ο Χαβιέ Νάρτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Αλγερία είναι μια χώρα με τεράστιους πόρους. Ωστόσο ε, η διακυβέρνηση είναι ολιγαρχική και διεφθαρμένη και υπόκειται ε, στον έλεγχο του ενός κόμματος που έχει όλες τις εξουσίες υπάρχουν, υπάρχει η νεαρή αλληλεγγύη, η οποία, υπάρχουν οι νέοι στην αλληλεγγύη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και της ανεργίας. Ο στρατηγός Αχμέντ Καϊτσάλαχ ε, ζήτησε να παραιτηθεί ο πλασματικός ε, ηγέτης ε, Μπουτεφλίκα ο, ο, η εξουσία ωστόσο θα παραμείνει στα χέρια του στρατού. Δεν θα πρέπει να, ε, να έχουμε καμία σύγχυση. Ε, ο στρατηγός ε, Σάλεθ με την υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού προετοιμάζει την μετάβαση. Το θέμα είναι ότι η διαφορά είναι ότι ο λαός ε, ξεκίνησε, άρχισε να εξεγείρεται και δημιουργήθηκε ωστόσο μία ψευδέστηση ότι ενδεχομένως θα υπάρξει μία αλλαγή ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ε, αποζητάει εξουσία να παραμείνει. Ε, ο στρατός θα πρέπει να καταλάβει ότι η εποχή της στρατηγικής εξουσίας έχει παρέλθει και θα πρέπει η κοινωνία να κάνει ένα άνοιγμα. Γιατί η Αλγερία βρίσκεται σε μια κομβική θέση ως προς την σταθερότητα της εποχής και είναι ανοιχτή προς, την, προς τις ώρες του Σαχέλ και προς την Μεσόγεια. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το λαό της Αλγερίας αυτή την αναγκαία μετάβαση. Θα πρέπει να να ε, συνειδητοποιήσουν ότι τους στηρίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον το οποίο θα σηματοδοτήσει μια θετικότερη εξέλιξη για όλους. Ευχαριστώ κύριε Νάρτα. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Φουρτασούν. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω όλους όσους βγήκαν στο δρόμο στην Ριελία με περήφανο τρόπο και υπήρχε και ηγεσία των γυναικών ε, τώρα ε, αυτοί που ε, εμπορεύονται το πετρέλαιο δεν μπορούν πλέον να εξουσιάσουν όμως για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι υπάρχει απόλυτη σιωπή και από την πλευρά των Βρυξελών, κύριε Επίτροπε, μεταξύ της Αδιαφορία και της παρέμβασης υπάρχει η ενδιάμεση οδός. Θα πρέπει να υποστηρίξετε με θουσιώδη και αδελφικό τρόπο το λαό της Αλγερίας. Θα πρέπει να ακούσετε τα αιτήματα του λαού της Αλγερίας και να υποστηρίξετε τα αιτήματα για δημοκρατία, για μια διακυβέρνηση που να βασίζεται στην αξιοπρέπεια και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπερασπίσουμε τους δρόμους των πόλεων της Αλγερίας για να υπάρχει δημοκρατική μετάβαση και να αποφύγουμε μια ψευδή ψευδή απλώς αντικατάσταση της σημερινή εξουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ουρτασούν. Ο Ουρμπάν Κρέσπο, εξ ονόματος της Γουέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι γυναίκες και οι άνδρες της Αλγερίας διαδηλώνουν στους δρόμους ε, γιατί έχουν κουραστεί από ένα ολοκληρωτικό ε, σύστημα εξουσίας ε, ο Μπουτεφλίκα ε, μετέφερε τις εκλογές και μίλησε για μια περίοδο μετάβασης. Όμως οι διαδηλωτές θέλουν πραγματική αλλαγή, μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που να καλέσει εκλογές και να τροποποιήσει το Σύνταγμα έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι ελευθερίες. Είναι μεγαλύτερες ειρηνικές διαδηλώσεις που έζησε η Αλγερία εδώ και χρόνια. Όμως είναι συντριπτική η διεθνή Η Αλγερία είναι ο τρίτος προμηθευτής αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τις πολυεθνικές πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει τους διαδηλωτές και τα αιτήματά τους εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στέλνουμε την υπερισπασή μας, ε, τη στήριξή μας στα αιτήματα μιας κοινωνίας ε, που ζητά δικαιοσύνη και δημοκρατία στην Αλγερία. Πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Ουρμπαν Κρέσπο. Ο κύριος Άρνοτ από το EFTD. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ τη σοβαρότητα της ε, κατάστασης στην Αλγερία. Οι διαδηλώσεις, ευτυχώς, μέχρι τώρα υπήρξαν ειρηνικές έχουμε διαδηλώσει με νέου που κατεβαίνουν στου δρόμου γιατί πιστεύουν ε, σε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσφέρει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Ένα από τα βασικά σχόλια που βλέπουμε ξανά και ξανά από τον κόσμο στην Αλγερία είναι ότι θέλουν οπωσδήποτε την ελευθερία έκφρασης. Να μπορούν λοιπόν να εκφραστούν με τρόπους που δεν μπορούσαν μέχρι τώρα. Όμως η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ε, είδαμε τον ε, στρατηγό σήμερα που ζήτησε ο Μπουτεφλίκα να ε, αποπεμφθεί ουσιαστικά, να θεωρηθεί ότι πλέον δεν μπορεί να ηγείται της χώρας. Όμως η ελευθερία έκφρασης θα πρέπει να συνδέεται και με την ανεξιθρησκεία που κατοχυρώνεται υπό το άρθρο 36 του Συντάγματος Αλγερίας που αναφέρεται ότι η ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων είναι απαράβατη. Όμως υπήρξε δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αλγερία και πιο συγκεκριμένα χριστιανικών μειονοτήτων, γιατί έχω συναντηθεί με πάστορες, δύο φορές μάλιστα, που ήρθαν στο Κοινοβούλιο για να μας μιλήσουν ε, για, για τα δεινά που περνούν αυτή τη στιγμή στην Αλγερία έχει περάσει από τη θέση 42 στη θέση 22 ε, στην κατάταξη ε, με τις χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη δίωξη των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων. Αντίστοιχα, έχουμε δει τι έχουν περάσει στην Αγγλικανική Εκκλησία της Αλγερίας όσοι προβάλλουν και προωθούν θρησκευτικά μηνύματα ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, ε, διώκονται και πολλέ άλλε κατηγορίε ανθρώπων που εκφράζουν τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει. Επομένω, σε όλε αυτέ τι περιπτώσει θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι χριστιανοί και άλλε θρησκευτικέ μειονότητε διώκονται στην Αλγερία τη στιγμή ε, που συζητούμε τέτοια πράγματα με τι επόμενε μέρε. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άρνοτ. Από το ΙΕΝΕΦ, e ο κύριο Ζακ Κολομιέ. Κυρία Πρόεδρε, ε, σε εποχές ε, γαλλικής κυριαρχίας η Αλγερία ήταν ε, παράδεισος, όχι πια όμως. Σήμερα, λοιπόν, αυτό γίνεται όλο ένα και πιο προφανές. Σε αυτό το ημικύκλιο που δεν είναι υπέρ μια ομαλή μετάβαση, αλλά τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τέτοια διαδικασία. Η Αλγερία δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όχι ακόμα. Επομένω, οτιδήποτε άπτεται τη Αλγερία ε, εναπόκειται στα χέρια των Αλγερινών. Αλλά βλέπουμε ότι οι ηγέτες τους ε, δεν μπορούν να την χειριστούν εδώ και 57 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λυθούν στην Αλγερία και πουθενά ε, βέβαια, ο Μπουτεφλίκα που έχει ε, πολλές φορές προσβάλει τους Γάλλους ε, δεν ε, μας δημιουργεί καμία αίσθηση συμπόνιας. Το μοναδικό λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι εξελίξει να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε αύξηση της μετανάστευση. Ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Κολεμπιέ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Αλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτρο. Εγώ παρακολούθησα τις τελευταίες εξελίξεις στην Αλγερία, την αναστολή των προεδρικών εκλογών, την ε, ζήτηση να απομακρυνθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι σημαντικό να γίνει η δημοκρατική μετάβαση η οποία να δώσει το λόγο στον λαό της Αλγερίας και να ανταποκριθεί στο αίτημα της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Να γίνει με μία μορφή που να μην ε, περιέλθει η χώρα αυτή στα, σε σφαλμένες ε, εμπειρίες που έζησαν οι γειτονικέ χώρες. Είναι σημαντικό με μία συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών να μπορέσουν να εκφραστούν όλες αυτές οι συλλογικότητες και με έναν αξιόπιστο τρόπο να ακουστεί η φωνή του αλγερικού λαού και να, δίνουν, ε, και να γίνουν ε, δίκαιες εκλογές. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να υποστηρίξει αυτές τις, ε, αυτό το αίτημα της ελευθερίας το οποίο ακούγεται όλο και περισσότερο στους δρόμους της χώρας αυτής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Αλγερία οι διαδηλώσει επαναλαμβάνονται συνεχώς. Είναι γιγάντιες ειρηνικές διαδηλώσεις και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι σκέφτεται η πλειοψηφία των Αλγερινών. Αρχικά οι διαδηλώσει ε, αφορούσαν την υπόθεση της πέμπτης ε, θητείας ε, του Μπουτεφλίκα. Τώρα ζητούν να κλείσει γρήγορα μεταβατική περίοδος. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν είναι να περάσουν από ένα έτοιμο εκλογών χωρίς τον Μπουτεφλίκα σε μια παραμονή του Μπουτεφλίκα χωρίς εκλογές. Γι' αυτό είναι απαραίτητο και εμείς να δείξουμε το δρόμο για μια λογική μετάβαση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο σταθερότητα στην Αλγερία, όπου η δημοκρατία και οι μεταρρυθμίσεις και τα δικαιώματα είναι ζωτικά. Το άρθρο 102 του συντάγματος ε, θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική της πολιτική να ασχοληθεί με αυτή τη χώρα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί αν ε, υπάρχει ισορροπημένη μεταβατική μετάβαση στην Αλγερία, εξαρτάται από αυτό το μέλλον όλη τη περιοχή. Ευχαριστούμε, κύριε Παντσιέρη. Ο Μαρέκ Γιούρεκ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, παρατηρούμε τα, τις εξελίξεις στην Αλγερία. Είναι απολύτως κατανοητό ότι η χώρα αυτή δεν βρίσκεται μόνο κοντά μας, αλλά έχουμε κατά νου τα όσα συνέβησαν την δεκαετία του 90, το τελευταίο δημοκρατικό πείραμα που οδήγησε στη νίκη του φιλελεύθερου μετόπου και στη συνέχεια ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος. Ε, και όλη αυτή η κρίση πέρασε και στην Ευρώπη. Και ε, παρόλο που είμαι αντίθετο προς την ε, Επιτροπή, θα πρέπει να αναγνωρίσω το γεγονός ότι ο κύριος Χάν με νυφαλιότητα παρατηρεί τις εξελίξεις στην ε, Αλγερία. Και πράγματι αυτό είναι εις όφελος της ε, προσυμφέρον της Ευρώπης. Ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα σφάλματα τα οποία διαπράξαμε στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες της ε, Αραβικής Άνοιξης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιούρεκ. Επόμενος ομιλητής, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σάιφη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Η καρδιά της Αλγερίας ε, ξαναρχίζει να πάλεται. Αυτό είναι από τα σλόγγαν που διαβάζουμε στους δρόμους της Αλγερίας εδώ και ένα μήνα. Θα ήθελα να ποτίσω τιμή στο λαό της Αλγερίας για το θάρρος του και την αποφασιστικότητα του. Η διοργάνωση ειρηνικών διαδηλώσεων υποδειγματική και αξίζει το θαυμασμό όλων μια κινητοποίηση όλων των γενεών και σε όλες τις περιοχές αξίζει κάτι περισσότερο από μια απλή ε, κυβερνητική ε, μεταρρύθμιση εκ μέρους της κυβέρνησης. Ε, η, χώρα έχει περιέλθει σε δινή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος αυτού του διακυβεύματος και να μην δώσει στο λαό της Αλγερίας την εντύπωση ότι δεν έχουμε κατανοήσει το βάθος των ετοιμάτων της. Το μέλλον μας ανήκει είναι ένα άλλο σλόγγαν, άλλο σύνθημα των ε, διαδηλωτών. Ο πληθυσμός Αλγερίας καταδεικνύει καθημερινά με αξιοπρέπεια και δύναμη ε, τον ε, αγώνα του για την ελευθερία και πραγματικά είναι ένα πολύ σωστό μήνυμα για την νεολαία. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λόπεθ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Σήμερα μιλάμε για την Αλγερία μετά από εβδομάδε ε, που κάθε Παρασκευή εκατομμύρια Αλγερινοί διαδηλώνουν εξωγηρημένοι για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στη χώρα. Ζητούσαν να μην υπάρξει η πέμπτη θητεία του Πρόεδρου